ξεκινάμε. Ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Παρακαλώ. ότι δεν έχω μαζί μου την ε, κάρτα την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, Δυστυχώ δεν την έχω μαζί μου, επαναλαμβάνω.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 θα διαρκέσει πολύ ψηφοφορία. Θα διαρκέσει ε, πολύ αυτή η ψηφοφορία. Και παρακαλώ λοιπόν, ε, αν μπορείτε να στείλετε κάποιον βοηθό σας να την ε, ψάξει αυτή την κάρτα, γιατί πολλά πολλά θα γίνουν. Ναι, έστειλα, έστειλα για να μου τη φέρουν. Μήπως χρειάζεται μερικά λεπτά για να σας δώσουν την κάρτα. Δεν ακούσαμε την απάντηση. Λουίς Δεμέρο, ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ η δουλειά σήμερα το πρωί. Ενώ λοιπόν περιμένει η κυρία τη ηλεκτρονική της κάρτα να ψηφίσουμε στην αρχή τουλάχιστον για να τάσω στις χειρός ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε ένα μέρος τουλάχιστον έτσι ναι θα ξεκινήσουμε αμέσω, λέει η πρόεδρος ψηφίζουμε λοιπόν την 242 τροπολογία ψηφίζουμε παρακαλώ Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 242. Ψηφίζουμε τώρα τη 243. Ψηφίζουμε. Chiusa la votazione. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 243. Ψηφίζουμε τη 244 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 245 ε, και ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται η 245. 246 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται η 246. 247. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται η 247. 2.48 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 318 ψηφίζουμε παρακαλώ. Όχι, ταυτόσημη. Άρα λοιπόν ψηφίζουμε την 2.49. Ψηφίζουμε για τη 2.49. Πέρας. απορρίπτεται. 250 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική λύση 1. Έχει ζητηθεί να ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Α. Παράγραφος. Το Calls on the Commission, ε, συνεργασία κλπ. μεταξύ των κρατών μελών. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος δεύτερο τμήμα να προσθεθούν για όχι διακόπτη η πρόεδρος τι έγινε καταπίπτει το δεύτερο τμήμα για τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Όχι, δεν καταπίπτει. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Στη συμβαστική λύση 1, σε δύο τμήματα και πάλι, να διαγραφούν ό,τι θα έπρεπε, να συμπεριλέγανε με στάλα κλπ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Να προσθεθούν τα ό,τι θα έπρεπε ανάμεσα στα υπόλοιπα, να συμπεριληφθεί κλπ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική λύση 2. Πρόταση 2. Ψηφίζουμε. Πέρας.

Ψηφίζουμε την 270. Παρακαλώ. Δεν ε, ψηφίζουμε ξανά γιατί είναι, έχει να κάνει με γλωσσική, με φραστική διατύπωση αυτό. Passiamo al 3 che pongo in votazione aperta. Ψηφίζουμε την συμβαστική 3. Chiusa la votazione. Approvato. Peras, engrinate. Την 272 ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 279. Ψηφίζουμε. εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 5 συμβαστική. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. ...284. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται. Τη 285 ψηφίζουμε τώρα. Παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται 285. 286 ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. 287 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 288 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 289 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 6. Συμβαστική 6 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Passiamo quindi al voto 298. Dichiaro aperta. 298 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρακόσια. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 626 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 301 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. δύο ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 303 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 304. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρία πέντε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 306. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 307. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 1308. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 309. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 310. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 311. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 312 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 313 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 314 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 315 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 317 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 316 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 329. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Συμβαστική 8 τι έχει. ότι είναι νόμιμο και όχι είτε νόμιμο και πρέπον. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 339. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. «340» και «341» ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε παρακαλώ τις δύο. Πέρας. Απορρίπτεται. 342. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική εννέα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 346. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 347, 348, δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέσσερα. 349 καταπίπτει. Η 350 τώρα ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 ψηφίζουμε. Πέρας. γκρίνεται Τρακόσια πενήντα ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. Τρακόσια εξήντα ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. για Σέντερο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πριν ψηφίσουμε το Συμβασμό 11 του κύριου Γιακολίνου, θα ήθελα να σας πω ότι η ομάδα μου ζήτησε το εξής. Επειδή θεωρούμε ότι υπάρχουν τροπολογίες που καλύπτονται από αυτό το Συμβασμό 395, 356, 398 και 442 που είναι μέτρα για την προστασία των θυμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο εισηγητής έλαβε υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις και την προστασία των θυμάτων, όμως στον συμβασμό απλώς τους κατονομάζει μέσα στα πλαίσια των συνόρων, της προστασίας των συνόρων. Εμείς θα θέλαμε να ψηφίσουμε ξεχωριστά αυτές τις ε, τέσσερις τροπολογίες που υποτίθεται ότι καλύπτονται από, από την τροπολογία συμβασμού, αλλά που στην ουσία δεν ε, καλύπτονται διότι δεν μιλάμε για την προστασία θυμάτων. Πρόκειται για τις 395, 97, 98, 442 που δεν καλύπτονται από την ε, πρώτα συμβασμού. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα Σέντερ. Η γραμματεία έχει λάβει αυτά τα δεδομένα, άρα θα ψηφίσουμε το συμβασμό και θα περάσουμε στις δικές σας τροπολογίες. 11. Ανοίγει η ψηφοφορία. Chiusa la votazione. Approvato. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα λοιπόν στην eh, ε, 374 που ψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. 374. Περνάμε στην 374, την οποία και ψηφίζουμε. Αυτή είναι μία... Ε, όχι, όχι, όχι, δεν είπα αυτή την... Ε, δεν ανέφερα αυτή την τροπολογία, κυρία Γιάλα Σέντερ. Ο εισηγητής θεώρησε ότι η 11 καλύπτει αυτές τις τροπολογίες. Δεν πρόκειται για τις επόμενες απλώς που μπορώ να δεχτώ. Δεν θα ήθελα όλες οι τροπολογίες να ψηφιστούν απλώς εκείνες που προβάλλουν την προστασία των θυμάτων, που είναι οι 395, 97, 98 και 442, που είναι πιο μετά στον κατάλογο ψηφοφοριών, που είναι τα συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των θυμάτων. Αυτές οι τέσσερις ε, για τις υπόλοιπες ε, δέχομαι τα δεδομένα. Δεν θα ήθελα να ψηφιστούν ξεχωριστά. Μόνο εκείνες που αφορούν την προστασία των θυμάτων. Θα ήθελα να ψηφιστούν ξεχωριστά. Ωραία, είναι σαφές. Περνάμε στο συμβασμό 12 που ψηφίζουμε. Τροπολογία συμβασμού 12. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία Συμβασμού 13. Ψηφίζουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 388. 388 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 388. 389. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε 490. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Το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 Τώρα ψηφίζουμε την 395, όπως ζήτησε η κυρία Γιάλα Σέντερ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 397. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 398. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Passiamo adesso, pongo in votazione il compromesso 14. Ψηφίζουμε την τροπολογία συμβασμού 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. 14. Πέρας. Εγκρίνεται. ψηφίζουμε την 403. Ε, Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία συμβασμού 15. Ψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 408. Αρχίζει η ψηφοφορία 408. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τις 409 ε, και 416 παρεμφερείς. Αρχίζει η ψηφοφορία επί των δύο. Πέρας. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε την 410. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ψηφίσατε όλοι, μπορούμε να κλείσουμε. Εγκρίνεται. 411. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 413. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Γυρνάμε λίγο πίσω, γιατί παρέλειψα την 412. Η 413 έχει εγκριθεί, τώρα ψηφίζουμε την 412. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται η 412. 415. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 417. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 418. Ε, 418 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 419. 419 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Τώρα ψηφίζουμε την 421. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 16. Ε, Ζητείτε ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Χωρίς τις λέξεις without, without the words suggest promoting the teaching. Ε, ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα αυτό. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Με την προσθήκη, με την προσθήκη του Transnational Cooperation. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 427. Ε, 427. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 428. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 429. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 17. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 434 ψηφίζουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. 434. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 434 πέρας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 435. Αρχίζει η ψηφοφορία. πέρας. Απορρίπτεται η 435.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 είναι 3,93, 3,90. Έχω την εντύπωση ότι τις περάσαμε χωρίς να τις ψηφίσουμε αυτές τις τρεις. Για ποιες λέτε. Έχουν εκπέσει αυτές οι τροπολογίες γιατί εγκρίναμε την τροπολογία συμβασμού. Γι' αυτό περάσαμε στην 434. Ψηφίζουμε την 436. Αρχίζει η ψηφοφορία. «436 πέρας». Εγκρίνεται. «437». 437 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 438. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 439 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 18. Ψηφίζουμε την τροπολογία συμβασμού. Όχι, με συγχωρείτε. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 441, μου λέει η γραμματεία. 441. Ψηφίζουμε. 441. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 18. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε την τροπολογία 442. 442. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 443. 443 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 444. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Τετρακόσα σαράντα επτά. Πέρας. ψηφίσουμε την 451. 451. Πρέπει να ψηφιστεί γιατί υπάρχει ασυμβατότητα με την άλλη. Θα πρέπει να δούμε ποια ε, έκδοση, ποια εκδοχή θα δεχτούμε.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 Devo porre in votazione l'emendamento. Ψηφίζουμε την 451. Είναι γλωσσικό το ζήτημα, αλλά επειδή υπάρχει ασυμβατότητα με τη δεύτερη τροπολογία, θα πρέπει να δούμε τι θα επιλέξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία 451. Πέρας για την 451 εγκρίνεται. Περνάμε στο συμβιβασμό 19. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 20. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία Συμβασμού 21. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία 468. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 469. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται.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 Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 472. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 474 Ζητείτε ξεχωριστή ψηφοφορία σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, όπου γίνεται μια προστίκη από το recommends μέχρι το bank. Ψηφίζουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε με την προσθήκη and business. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και το τελευταίο κομμάτι. Calls on member state uh, on procurement. Ψηφίζουμε. η ψηφοφορίας. Τέλος. Το τρίτο τμήμα απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε... Α, ο κύριος Μπορσέλη. Sì, volevo proporre un emendamento orale al 475. Να βγάλουμε αυτό το καθοριστικό, να το αφαιρέσουμε σαν λέξη. Έτσι. Κάποια αντίρρηση πάνω στην παρουσίαση αυτής της προφορικής τροπολογίας. Κοιτάξτε, μα έχουμε ήδη ψηφίσει γι' αυτό. Δεν μπορούμε ε, να ψηφίσουμε, να αποφασίσουμε για κάτι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. 475. Συγγνώμη, στην 475 ζήτησε την προφορική ερώτηση προχωράμε με την αλλαγή αυτή. Ψηφίζουμε λίγο. Λοιπόν. Votazione conclusa. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 485. Ψηφίζουμε. Τέλος. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 485. 486. 486. Τέλος. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την συμβαστική 23. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 495. Ψηφίζουμε. 495. Γύρω γύρω του είναι γυναίκες, γεμάτο γυναίκες και τον κάνουν και αφαιρείται. Τέλος της ψηφοφορίας. 496 ψηφίζουμε. Τέλος. εγκρίνεται. Η επόμενη 497 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Και τώρα την 498 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 499 αρχή της ψηφοφορίας τέλος εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε την 500 τροπολογία 500 αρχή της ψηφοφορίας τέλος απορρίπτεται. 501 ξεχωριστή ψηφοφορία έχει ζητηθεί. Το πρώτο κομμάτι ψηφίζουμε. Ξεκινάμε με το support Training. Αρχή της ψηφοφορίας για το πρώτο τμήμα της 501. Τέλος. Εγκρίνεται. Και τώρα το δεύτερο τμήμα. Προσθέτουμε Independent Advice for Civil Servants, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Και τώρα περνάμε στην 503. 503, αρχή της ψηφοφορίας. «503, τέλος της ψηφοφορίας». Απορρίπτεται η 503. Και τώρα ψηφίζουμε την 504. 504, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην συμβιβαστική 24 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται περνάμε κατευθείαν στην συμβιβαστική 25. Ψηφίζουμε την 25, αρχή της ψηφοφορίας. Συμβιβαστική 25. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην συμβιβαστική 26. Ψηφίζουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβιβαστική 27, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 521. 521. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην συμβιβαστική 28. Αρχή της ψηφοφορίας. Συμβιβαστική 28. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29. Ψηφίζουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 537. Ψηφίζουμε. 5-3-7. Ε, 6, συγγνώμη, 5-3-6. Πέρας. Απορρίπτεται η 536. Και τώρα ψηφίζουμε την 537. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίσουμε την 538 και την 539 μαζί. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική 33. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Η 33 εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 30, συμβιβαστική 30, αρχή της ψηφοφορίας. 30, συμβιβαστική τροπολογία 30. Πέρας. εγκρίνεται. Και περνάμε στην 548. Ψηφίζουμε την 548. Αρχή. 548 ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 549, αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την 550. 550. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 551. 551. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 552. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την 553, αρχή της ψηφοφορίας. 553. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32. Ψηφίζουμε. Πέρας. Συμβιβαστική 32. Και τώρα ψηφίζουμε την 572. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε συμβαστική 34. και εδώ υπάρχει ξεχωριστή ψηφοφορία, το πρώτο τμήμα, offering μέχρι offense. Αυτό είναι το κομμάτι το πρώτο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο κομμάτι που είναι ότι προσθέτουμε offering μέχρι offense. Ναι. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, όχι. Ψηφίζουμε το δεύτερο κομμάτι Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την 581. 581, αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την συμβιβαστική 36. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 36 Πέρας. Η 36 εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την 592. Ψηφίζουμε την 592. Πέρας. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην επόμενη, 593, αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στη συμβαστική 37. Αρχή της ψηφοφορίας, συμβιβαστική 37. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 596. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 597. Ψηφίζουμε. πέρας. Η 597 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 598. Πέρας. Απορρίπτεται. 599. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 38. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. εγκρίνεται. Περνάμε στην 604. Αρχή της ψηφοφορίας. 604. 604. Πέρας. Απορρίπτεται. 39. Συμβιβαστική 39. Αρχή της ψηφοφορίας. 610 ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την 610, αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Και τώρα περνάμε στην 618. 618. Πέρας. 618. 618. Πέρας. Υπάρχει πρόβλημα ναι, το βρήκατε. Ψηφίσατε. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την συμβιβαστική 40. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 41, συμβιβαστική 41, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 42, συμβιβαστική 42. Ψηφίζουμε. Τέλος. εγκρίνεται και περνάμε στην 624. 624. Θέλω να αποσύρω αυτή την τροπολογία, Πρόεδρε. Ωραία. Άρα περνάμε στην 6.30. 6.30 ψηφίζουμε. 630. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την 635, αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 636. 636. Απορρίπτε. Ω, έχει αποσυρθεί. 6.37. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 636. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 639. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. εγκρίνεται. 6.40 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβιβαστική 43, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται η 43. 643. Ψηφίζουμε παρακαλώ την 643. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 44. Σε δύο τμήματα η ψηφοφορία αυτή. Έτσι έχει ζητηθεί. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα για τις εθνικές αρχές κλπ. κλπ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο μέρος, δεύτερο τμήμα. Μέχρι τον προστατευτικό μηχανισμό. Αυτό να προσθεθεί. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται 648 ψηφίζουμε 648 Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται 649 ψηφίζουμε Πέρας. Εγκρίνεται. 650. Ψηφίζουμε. 650 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 651 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 652 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 653 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 654 ψηφίζουμε. 654. πέρας είπαμε. 654. Απορρίπτεται. Ο κύριος Κυλακάκης μήπως θα ήθελε κάτι να πει. Όχι. Απορρίφθηκε η 654. 655 τώρα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 656. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 657 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 45 συμβαστική 45 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται Συμβαστική 46. Ψηφίζουμε 46. Πέρας. Εγκρίνεται. 668. Ψηφίζουμε. 668. Πέρας. εγκρίνεται. 669 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε. 700, μάλλον 670 ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται. 771 υπέρ, ε, συγγνώμη, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 672. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. 673 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 674 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Μποσκού δεν ψηφίσαμε την 663 και 664, αν δεν κάνω λάθος. Τις παραλείψαμε. No, but it falls, it falls till 662. Μέχρι το 662 ε, αλλά η 663 και 664 δεν εντάσσονται στο συμβιβασμό, στην πρόταση συμβιβασμού. Έχετε δίκιο, κύριε Μποσκούρ. Και την 663 και την 664 πρέπει να τις ψηφίζουμε. Την 663 ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 664. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται που είχαμε μείνει ξεκινάμε πάλι από εκεί κύριε Μποσκού ευχαριστούμε 675 ψηφίζουμε την 675 πέρας εγκρίνεται 676 ψηφίζουμε. Πέρας. Σαρανταεφτά συμβαστική ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 682 Ψηφίζουμε. 682. Πέρας. Εγκρίνεται. 683 ψηφίζουμε. Πέρας. Συμβαστική 48. Πέρας. Εγκρίνεται. 687. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 49. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 695. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες 696-697. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Και δύο ακόμα. Ταυτόσημες τις ψηφίζουμε 698, 699, ψηφίζουμε τις δύο, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική 50, όχι, η 700, ψηφίζουμε την 700 τελικά. Τροπολογία 700. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 50. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την 50. Συμβαστική. Πέρας. Εγκρίνεται. 706 ψηφίζουμε την 706. Πέρας. Εγκρίνονται. 709 ψηφίζουμε. 709 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 710 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 711 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 712 ψηφίζουμε. σκέφτεται 713 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 714 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 7-16 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 7-17 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 718 Ψηφίζουμε. Πέρας. Επτά δεκαεννέα. Ψηφίζουμε. Πενήντα ένα συμβαστική. Ψηφίζουμε παρακαλώ. 728. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 729 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 7.31 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 7.32 ψηφίζουμε. Πέρας. Επτά Εγκρίθηκε 732. Ψηφίζουμε λοιπόν την 733. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 734 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 735 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 736 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 737 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 738. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 739. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 7.40 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 7.42 ψηφίζουμε. 7.42. Πέρας. Απορρίπτεται. 743 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 744 ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτεται. Και τροπολογία 1 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Οι 2 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ψηφίζουμε. 4 είπαμε. 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Καταπίπτει η 5. Η 6 τώρα. Ψηφίζουμε για την 6. Πέρας. Εγκρίνεται. 7 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται η 7, 8 τώρα. Ψηφίζουμε για την 8. Πέρας εγκρίνεται. 9. Ναι, Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 11 τώρα. Ψηφίζουμε. 11 πέρας εγκρίνεται 12 ψηφίζουμε πέρας Approvato, pongo in votazione l'emendamento 13 ψηφίζουμε Πέρας. Δεκατρία. Απορρίπτεται. Δεκατέσσερα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκαπέντε. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. 16 ψηφίζουμε. 16 είπαμε. 60 αν το θέλετε και αγγλικά. 16, 16 συγγνώμη. Εγκρίνεται. 17 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 18. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 19. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, αποσύρω την 20 διότι δεν συμμετεί με την 9. Σας ευχαριστούμε κύριε Μίσελ. 21 τώρα. Ψηφίζουμε την 21. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 23. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. 25. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 26. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 ψηφίζουμε τροπολογία 27 πέρας εγκρίνεται 28 ψηφίζουμε εγκρίνεται Δεν δεχόμαστε το 29, άρα λοιπόν δεν το ψηφίζουμε. Την 30 τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 32. Τροπολογία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 52. Ψηφίζουμε. Πέρας. 53 συμβιβαστική. Ψηφίζουμε. Πέρας της Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Ψηφίζουμε. 38 είπαμε. Πέρας. Εγκρίνεται η 49 τώρα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 54 τροπολογία. 54. Ψηφίζουμε. Πέρας. 54 είπαμε κύριε Μίτσελ. Εγκρίνεται. 43 Ψηφίζουμε. 43. Πέρας. Απορρίπτεται. 55. Ψηφίζουμε. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 52. ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται στη 53 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα να αφαιρεθεί μέχρι το οικονομική ανάπτυξη Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα της 53. Να προσθέσουμε μέχρι και πάλι το κομμάτι αυτό το οικονομική ανάπτυξη. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται 56 συμβαστική ψηφίζουμε πέρασε εγκρίνεται 57 ψηφίζουμε πέρας 57 είπαμε Συμβιβαστική. Εγκρίνεται. Εξήντα τροπολογία. Ψηφίζουμε. Εξήντα ένα. Πέρας. Εγκρίνεται. 62 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 63 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 64 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 65. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 66. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 58. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 59. Συμβαστική. Ψηφίζουμε. 59. Συμβαστική. Πέρασε. εγκρίνεται. ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 80. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται 81 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 82 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 83 ψηφίζουμε Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 60. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Ψηφίζουμε. Α, λεπτό. Ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται 92 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 93 ψηφίζουμε πέρας Respinto. Απορρίπτεται. Συμβασμός 61. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 100. Ψηφίζουμε την τροπολογία 100. Ψηφίζουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 101. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 102. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 62. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 63. Ψηφίζουμε το συμβιβασμό 63. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 64. Ζητείτε ξεχωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, χωρίς τη λέξη terrorism. Αρχίζει η ψηφοφορία, χωρίς τη λέξη terrorism, πέρας, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα της 64 όπου προστίθεται η λέξη terrorism. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 121. Ψηφίζουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. 121 ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. 122. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 123. Αρχίζει η ψηφοφορία. 123. Πέρας. Απορρίπτεται. 65. Αρχίζει η ψηφοφορία. 65. Πέρας. Ψηφίσαμε την 65. Συμβασμός 65. Εγκρίνεται. 127. Ψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία 127 πέρας εγκρίνεται συμβιβασμός 66 66 ψηφίζουμε πέρας περνάμε στην 135. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 135. 136. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 7. Συμβασμός 67. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 140. Ψηφίζουμε την 140. Πέρας. Εγκρίνεται ψηφίζουμε το συμβασμό 68. 68 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 149. Ψηφίζουμε. 149. Πέρας. εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το συμβασμό 69. 69 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 159. Ψηφίζουμε από κοινού δύο παρόμοιες τροπολογίες, 158 και 159 και 160. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Ψηφίζουμε την τροπολογία. Καταπίπτει 161. Περνάμε λοιπόν στο συμβασμό 70. Αρχίζει η ψηφοφορία 70. Πέρας. 165 ψηφίζουμε. Εκατόν εξήντα πέντε ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. Passiamo al compromesso Συμβασμός 71. Ζητείτε ξεχωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα όπου βγαίνει το online trafficking in the creative content. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα του Συμβασμού 71, όπου προσθέτουμε τις λέξεις online trafficking in creative content. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 177. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 178 προφορική. Κανείς δεν αντιτίθεται νομίζω. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική η οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 72. Συμβασμός 72. 72. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 185. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 186 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 187 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 188 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 189 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 73 Συμβασμός 73 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 193. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 194 αρχίζει η ψηφοφορία. 194. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 74. Συμβασμός 74 ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται. 204-205 παρόμοιες, παρεμφερείς, αρχίζει η ψηφοφορία. 204-205 πέρας, εγκρίνονται. 206 αρχίζει η ψηφοφορία. 206 πέρας, εγκρίνεται. 75. Συμβασμός 75. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε δύο πανομοιότυπες, τη 211 και 12. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 213 ψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 76, συμβασμός 76, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Επί της 76 εγκρίνεται. εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στον συμβιβασμό 77. 77 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 230 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 231. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 232. Αρχίζει. Πέρας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 233. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 234. 234. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 235, 235. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 236. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 237. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 238 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 239. Πέρας. απορρίπτεται. 240 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 241. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 241. πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα θα ήθελα... Stop, stop, stop. Θα ήθελα να ψηφίσουμε την πρόταση ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Με 24 ψήφους υπέρ και 5 αποχές, κανείς δεν ψήφισε κατά, εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια κύριε Γιακολίνο, θέλετε να παρέμβετε, έχετε το λόγο εντάχει, γιατί φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι είναι κουρασμένοι όσο και εσείς και εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στη γραμματεία, του συμβούλους που συνεισέφεραν και εσάς για μια εργασία η οποία ήταν ποιοτικά πολύ καλή και ε, καταπολεμά το οργανωμένο έγκλημα και τις ε, δραστηριότητες ε, τύπου μαφίας. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Σήμερα στις 3 θα αρχίσουν στις εργασίες μας με τα κοινοβούλια των άλλων κρατών μελών. Ο κύριος Νιούτον Ντάν ζήτησε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε εσάς για τον τρόπο με τον οποίο έχετε καθοδηγήσει και δεκτάει την αποτελεσματικότητα της τροπολογία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Με βοήθησε η εξαιρετική γραμματεία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους.